was 2.56 on that clock. Good morning, colleagues. I'm sorry for the late... Καλημέρα, συνάδελφοι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Sorry. Oh, you wanted to talk to uh, Claudia. Okay, that's fine. That is also important. So let's um, begin. I'm sorry. Ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη που αργήσαμε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας γίνεται συνεδρία σε ένα ψηφοφοριών. Την ψηφοφορία την κάναμε αρχές εβδομάδας, διότι το ΕΛΚ έχουν σήμερα συνεδρίαση στο Ελσίνκι. Θα έχουμε την επόμενη Πέμπτη στο Στρασβούργο σύντομε ψηφοφορίε. Έπρεπε να κάνουμε ανακατατάξει. Συγγνώμη κύριε πρέπει ξεκινάμε το σημείο σα λίγο αργότερα. Ξεκινάμε λοιπόν. Με την έγκριση μερίσια διάταξη θεωρείται συγκεκριμένη. Γλωσσική γλωσσικό συνδυασμό έχουμε εκτό από κρατικά, δανέζικα, μαλτέζικα, ουγγρικά, γοδελικά. Έχουμε όλε τι γλώσσε. Πάμε στο σημείο του κυρίου Ντιπχέ. Εξετάζουμε τροπολογίε όσον αφορά την έκθεση του. Η ενίσχυση τη ασφάλεια των ταυτοτήτων της, των πολιτών τη Ένωση. 205 τροπολογίε έχουμε. Και έχουμε γνωμοδότηση τη Επιτροπή Γυναικών Συνεδρίαση, συνεδρίαση ανεσκιώδης ήδη πέντε φορές. Έγινε σκληρή δουλειά. Αμιλητή θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντιπρέ για να μας βγαίνει η κατάσταση. Ζεράρ, έχεις το λόγο. Α, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Έκαναν προσπάθεια να είναι εδώ σήμερα. Να υπενθυμίσω το στόχο της πρότασης. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις ταυτότητες εθνικές από ευρωπαϊκή. Να είναι σαφές. Και να μην υποχρεώσουμε τις χώρες που δεν έχουν ταυτότητα να εκδώσουν ταυτότητα. Θέλουμε μόνο να ισχύσουμε τα στοιχεία ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των ταυτοτήτων και των αδειών διαμονής που εκδίδονται από τα κάτι μέλη. Στόχος σαφέστατος. Να ευνοήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών ελαχιστοποιώνταν στον ελάχιστο βαθμό τη δυνατότητα πλαστογράφησης και κατάχρησης ταυτότητας. Η πρωτοβουλία είναι απαραίτητη. Να υπενθυμίσω, 250 διαφορετικές εκδοχές έχουμε δελτίων ταυτότητας ή αδειών διαμονής στην Ένωση. Δελτία ταυτότητας, άδεια διαμονής, των οποίων το επίπεδο ασφαλείας ποικίλει και σημαντικά. Γι' αυτό Υποστηρίζω, όπως και πολλοί εμπειρογνώμονες και όπως προβλέπεται στην πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υποχρεωτική εγγραφή δύο στοιχείων βιομετρικών, δαχτυλικών αποτυπωμάτων και προσώπου στις τυποποιημένες πλέον ε, ταυτότητες. Όσον αφορά τόσο ευαίσθητα στοιχεία όπως τα δαχτυλικά αποτυπώματα, είναι απαραίτητο να προβλέπονται τα αναγκαία χέγγια που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Χρειάζονται και άλλα χέγγια όσον αφορά την ε, εισαγωγή των στοιχείων, κυρίως όσον αφορά τα παιδιά ή ευάλωτα άτομα. Ότι τα παιδιά να μην υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση παρά μόνο από την ηλικία των 12 ετών. Τρίτον, τα δαχτυλικά αποτυπώματα που θα λαμβάνονται θα αποθηκεύονται μόνο για την αναγκαία περίοδο για να μπουν στο τσιπάκι πριν να σβήσουν. Τέταρτον, ότι η προτινόμενη διατάξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν νομική βάση, ούτε να δημιουργηθεί ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ταυτοτήτων, ούτε να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων εθνικές, που αυτές μόνο μέσω των νομοθεσιών των κρατών μελών μπορεί να δημιουργηθούν. Πέμπτον, η πρόσβαση στα βιομετρικά στοιχεία να περιορίζεται αυστηρά στο προσωπικό των αρχών των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένα με την ταυτοποίηση των ατόμων. Να υπενθυμίσω προφανώς ότι χρειάζεται σωστή ε, προσέγγιση και να υπάρχουν τα αναγκαία χέγγια όταν τα κράτη-μέλη ε, δίνουν σε υπεργολαβία την έξοδο ταυτοτήτων. Υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Έχω και διάφορες άλλες προτάσεις πέραν των βασικών για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, κυρίως μέσω αναγκαίας ανταλλαγής, ε, ανταλλαγής κλειδών ε, αποκρυπτογράφηση. Η, εφαρμο, η αμοιβαία αναγνώριση των προσωρινών ταυτοτήτων, η περίοδο συλλογής των στοιχείων και η ευρωπαϊκή σημαία να πηγαίνει πάνω από τις εθνικές σημαίες όσον αφορά τα έγγραφα αυτά των ταυτοτήτων. Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως υπενθυμίσατε κύριε Πρόεδρε, ήδη τα συζητήσαμε. Ανταλλάξαμε απόψεις σε πέντε συνεδρία και οδών και θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τις εκφραστήσεις απόψεις των ομάδων. Αυτές οι προσπάθειες και οι συνομιλίες έλαβαν χώρα και θα λάβουν χώρα, ελπίζω, σε έξοχο κλίμα και ευχαριστώ δημοσία του συναδέλφου των άλλων ομάδων, τους συνεργάτες τους και τη γραμματεία της Επιτροπής μας. Δεν αφισβητώ ότι μέσω αυτών των συζητήσεων και από τη βούληση της συμφιλιώσεως και για το κοινό καλό των Ευρωπαίων πολιτών θα καταλήξουμε προσεχώς σε μια συμφωνία που θα τύχει ευρεία υποστηρίξεω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, με ανυπομονησία και ενδιαφέρον και με ηρεμία και γαλήνη περιμένω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ζεράρ. Πάμε στους Κιώδης τώρα. Ιώσεφ Ρενεχόλτσερ, που αντικαθιστά την Σιλβή Φων Κάουφμαν. Ζώσεφ, έχεις το λόγο. Η ε, κυρία Κάφμαν, η η εισηγήτρια, λοιπόν, ήθελε να μεταφέρει το εξή ε, μήνυμα. Δυστυχώ δεν μπορεί να παραβρεθεί σήμερα και έτσι Θέλει παρόλα να εκφράσει κάποιες ε, σκέψεις, να ευχαριστήσει καταρχάς ε, τον εισηγητή και για την δουλειά που έκανε και για την επικοδομητική συνεργασία. Θα ήθελα να επισημάνει δύο στοιχεία, καταρχάς ότι υπέβαλε τροπολογίες ε, καταρχάς. Πέρα από την απέτηση για την λήψη διπλού αποτυπώματος, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση αυτή. Η οποία όμως η κυρία Κόφμαν θεωρεί ότι αποτελεί παραβίωση για τα δικαιώματα των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό θα άγγισε πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δυσανάλογο ως μέτρο και δεν υπάρχει επίσης και ουσιαστική δικαιολογία, ουσιαστικός λόγος για να γίνεται αυτή η λήψη. Γι' αυτό λοιπόν ε, έχει υποβάλει η τροπολογία να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ε, και στο μέλλον τι ακριβώς θα κάνουν και πώς θα αλλάξουν, αν αλλάξουν τη σχετική τροπολογία. Υπέβαλε λοιπόν σχετική τροπολογία η κυρία Κάουφμαν σε ό,τι αφορά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και αυτό συνάδει και με αυτά που ζητάει ε, ο Ευρωπαίος Συνταλμένος για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων. Είναι μια δεύτερη τροπολογία για ε, τις αυτοτήτε που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας. Ε, θεωρεί ότι καλά θα ήταν να υπάρχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, να προβλέπεται μεγαλύτερη χρονική περίοδο δηλαδή. Και προ την κατεύθυνση αυτή κατέθεσε σχετικέ τροπολογίε. Θα πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία μέχρι την διάρκεια ισχύω του ε, γράφου. Προσβλέπει τη μελλοντική συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές, η κυρία Κάφμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος και οι σκιώδης από το ECR. Ο κύριο Βεστεσέν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους όλους. Τι να πω, ότι ο εισηγητής ε, έκανε μία πρώτη απόπειρα να βρει συμβιβασμού μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Γενικά είμαι ικανοποιημένο με το πώ πάνε οι τροπολογίε ε, και οι διαπραγματεύσει ε, ω τώρα. Και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παραστώ στι συνεδριάσει των σκιωδών. Έστειλα φυσικά του συμβούλου μου και με ενημέρωσαν σε ό,τι αφορά του βιομετρικού δείκτε. Αντίθετα με τι απαιτήσει κάποιων πολιτικών ομάδων για το ECR, είναι βασικό το ζήτημα του να υπάρχουν αυτοί οι δύο δείκτε επίση ό,τι αφορά τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, πιστεύουμε ότι η καλύτερη θέση θα ήταν να μείνουμε στα έξι χρόνια, γιατί εκεί μπορούμε να αποδείξουμε την αξιοπιστία των δακτυλικών αποτυπωμάτων και ότι αυτό συνάδει και με την πρόταση του VIS. Και σε ό,τι αφορά τι διατάξει ε, τη Eurocast, ε, του κανονισμού και τη αναθεώρηση αυτό. Τέλο, είναι σημαντικό για μα ε, το ότι υπάρχει αυτή η απόφαση να, ε, να δημιουργηθεί μια εθνική βάση δεδομένων, ένα εθνικό μητρό τεχνικών απομάτων, αλλά αυτό να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Και γενικά προσβλέπουμε στη συνέχεια τη συνεργασία με τον εισηγητή προκειμένου να βρούμε τι κατάλληλε και δέουσε λύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα, λέει ο πρόεδρο, η Σιλβί Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση στον Ζεράρ Ντεπρέ για το θέμα της ηλικία. Σε αυτά που είπατε, άκουσα, μιλούσατε για 12 ετών. Σε άλλα κείμενα, η ελάχιστη ηλικία δεν είναι αυτή. Τελικά, τι προέχει θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι και με τα υπόλοιπα κείμενα, δεν έχει σημασία. Τι ισχύει. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Σοφή, και πριν επανέλθουμε στον εισηγητή, να δούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, θέλω κι εγώ να τονίσω του στόχου, όπως έκανε και ο συγητή. Πρώτον, να διευκολύνουμε την ελεύθερη διακίνηση και δεύτερον, ελεύθερη κυκλοφορία και δεύτερον, να μπορούν οι πολίτες να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό πρόσκοπτα. Γι' αυτό εισάγουμε και το θέμα των δακτυλικών ε, αποτυπωμάτων. Διευκρινίζουμε ότι αν δώσουμε περισσότερη σημασία στην ασφάλεια, τότε δικαιολογείται στο τσίπ να έχουμε και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Δεν πρόκειται εδώ για την νομική βάση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων για δακτυλικά αποτυπώματα. Αν θέλουν μια τέτοια βάση δεδομένων οι ευρωβουλευτές για τα δακτυλικά αποτυπώματα, αυτό απαιτεί εθνική νομοθεσία και η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να συμμορφώνεται βέβαια με ε, τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων. Όσον αφορά την ηλικία, η Επιτροπή πρότεινε να παίρνουμε δακτυλικά αποτυπώματα από την ηλικία των 12 ετών και μετά, γιατί βασιζόμαστε ε, στον κανονισμό για τα διαβατήρια. Πράγματι, κάποια κείμενα μιλάνε για νωρίτερα. Εμείς θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε με τις ταυτότητες και με τα διαβατήρια. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητέ για τις συναντήσεις όπου είχαμε την δυνατότητα και εμείς να εξηγήσουμε τις ε, τεχνικές πτυχές του φακέλου αυτού. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη συνεργασία. Πρόεδρος, μάλιστα, επιστρέφουμε στον κύριο Ντεπρέ για να απαντήσει και να κλείσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέρφους που πήραν το λόγο εδώ. Όσον αφορά την θέση που ακούσαμε εκ μέρους τη Σιλβί Κάφμαν, ε, τη γνωρίζουμε και όντω αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της συζήτησης που πρέπει να κάνουμε για να αποφασίσουμε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο είναι αναγκαίο να έχουμε τέτοια δεδομένα, δακτυλικά αποτυπώματα δηλαδή, για να εξασφαλίσουμε περισσότερη προστασία από τα έγγραφα αυτά ταυτότητας. Είχαμε διάφορες συναντήσεις σκιωδών και ακούσαμε τα όρια. Τα όρια τα οποία γίνονται όλο και μεγαλύτερα όσο προχωράει η τεχνολογία. Δηλαδή ότι μόνο η φωτογραφία του προσώπου δεν φτάνει για να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται όντω για το συγκεκριμένο άτομο. Δεν θα σας μιλήσω εγώ για τις τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά μας εξήγησαν ότι η ταυτοποίηση του ατόμου μόνο βάσει της φωτογραφίας του ατόμου δεν φτάνει ότι η τεχνολογία επιτρέπει να παρέμβουμε στη φωτογραφία αυτή και να υπάρξουν έτσι απάτες. Οπότε πέρα από την φωτογραφία του προσώπου χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία. Ξέρω όμως ότι είναι ένα από τα πιο λεπτά ζητήματα και δύσκολα στις διαπραγματεύσεις αυτές που θα έχουμε για να αποφασίσουμε. Όσον αφορά τώρα την προβληματική της προθεσμίας για την εφαρμογή του μέτρου, καταλαβαίνω τα επιχειρήματα της κυρίας Κάφμεν που μας παρουσίασε ο συνάδελφος. Εδώ πέρα πρόκειται για μια διεύρυνση κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην φτάσουμε κάποια στιγμή οι χώρες ε, μέλη να πνιγούν, να έχουν ε, εκατομμύρια αιτήσει για αλλαγή ταυτότητας και να υπάρξει στραγγαλισμός γιατί δεν θα τα καταφέρνουν. Αυτά μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Βίστησεν για το θέμα. Τώρα κύριε Βίστησεν επίσης για, το... για αυτό που ζητάτε, δηλαδή η απόφαση για τη δημιουργία βάσης δεδομένων όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα να είναι εθνική αρμοδιότητα είναι σαφές. Από τη μια μεριά έχουμε την πρόταση πάνω στην οποία δουλεύουμε που είπαμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει νομική βάση αυτή καθεαυτή για να δημιουργηθούν εθνικές βάσεις δεδομένων αλλά από την άλλη οι χώρες μέλη εφόσον το επιθυμούν μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες βάσεις δεδομένων από το νομικό του σύστημα. Για την ηλικία, για να απαντήσω τώρα και στη Σιλβίκη Γιώμ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε και είπε ότι η ηλικία αυτή είναι η ηλικία που έχουμε προκειμένου να παίρνουμε δακτυλικά αποτυπώματα για τα διαβατήρια. Και το κάνω και εγώ για να συμφιλίωσω κάπως τις απόψεις. Είναι από τα θέματα που θα πρέπει να αποφασίσουμε στη συνέχεια, γιατί κάποιες ομάδες θεωρούν ότι η ηλικία από την οποία μπορούμε να παίρνουμε δακτυλικά αποτυπώματα είναι τα έξι χρόνια και άλλοι λένε στα 14 μόνο. Οπότε λαμβάνοντα υπόψη μα ότι υπάρχει το προηγούμενο των διαβατηρίων, ότι οι θέσει διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ του, προσπάθησα να καταλήξω σε μια ηλικία που να δικαιολογείται. Πρώτον, γιατί υπάρχει κάποιο προηγούμενο και δεύτερον, γιατί αποτελεί ένα σεβασμό που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι αποδεκτός δεδομένης της σημερινής κατάστασης. Αυτά, Πρόεδρε, είχα να πω και είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχίσουμε την συνεργασία μας σε πνεύμα συνεργασίας για την εξέβρεση συμβασμού και ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία σύντομα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεπρέ, λέει ο Πρόεδρος. Ή 3 ή δέκα του μηνός θα ψηφίσουμε. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα. Σας ευχαριστώ πάντως για την παρουσία σας εδώ και σας και τους κοιόδης συγητές. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο σημείο 4. Εδώ έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ε, τη στάκτη για την εφαρμογή των διατάξεων των συνθηκών σχετικά με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται στα άρθρα 2 και 6 της Εθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άτομο είναι στο κέντρο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου. Το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης της κυρίας ε, Άντερσον εξετάζει κατά πόσο οι διατάξεις των συνδικών είναι αρκετά αποτελεσματικές και θα κάνει κάποιες συστάσεις στις χώρες μέλη και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εξετάζει διάφορε πτυχέ που συνδέονται με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τα πολιτικά δικαιώματα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην Μαρτίνα για την γνωμοδότηση αυτή. Έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι θα συμφωνούν ότι λόγω του αριθμού λέξεων που επιτρέπονται σε κάθε γνωμοδότηση, οδήποτε αρχικό κείμενο γνωμοδοτήσεως μπορεί να περιέχει μόνο ένα κείμενο συγκεκριμένου όγκου. Η μόνη δυνατότητα να επεκταθούμε είναι μέσω τροπολογιών. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσω τις τροπολογίες για να βελτιώσω τη διατύπωση και να αποσαφηνίσουμε κάποια σημεία. Και ενθαρρύνουν συναδέλφους να συνεργαστούν μαζί μου. γνωμοδότηση διανεμήθη για να τη διαβάσουν τα μέλη. Είναι ένα πρωτόλιο το κείμενο. Μετά από συνομιλίες έθεσα προτεραιότητες. Να προστατεύσω όλα τα δικαιώματα, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, δημοκρατικά, περιβαλλοντικά. Δικαιώματα που συνδέονται με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για όλους τους πολίτες των κρατών μελών. Η προστασία των πολιτών στο επίκεντρο της προσπάθειας. Θα υποβάλουμε κάποιε τροπολογίες για να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή. Εκπροσώπηση των δικαιωμάτων ψηφού είναι κάτι σημαντικό πολιτικά δικαιώματα. Χρειάζεται να υποβληθούν τροπολογίες ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη το άρθρο 22 της ε, συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του 10 για της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δικαίωμα που στις εκλογές που περιγράφει ε, τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα δικαιώματά τους, όπως είπαμε, στο επίκεντρο του εγχειρήματο. Θα ήθελα να συνεργαστούν οι σκιώδεις για τυχόν τροπολογίες. Αναγνώριση αξίας και τη σημασία χάρτα των μελιδών δικαιωμάτων είναι κάτι που αναφέρεται στη γνωμοδότηση. Θέλουμε να το υποστηρίξουμε περαιτέρω. Και ότι έχουμε 1,8 εκατομμύρια πολίτε τη Ευρωπαϊκή στη Βόρεια Ιρλανδία και λαμβάνοντα υπόψη αυτά που υπόθηκαν το Δεκέμβριο του 2017 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι 1,8 εκατομμύρια πολίτε θα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά του και έχουν πρόσβαση εκεί που διαμένουν στα πολιτικά δικαιώματα. Μια τέτοια γνωμοδότηση είναι μια ευαίσθητη, αποτελεί μια ευαίσθητη ισορροπία. Προσπαθεί να καλύψει πολλά σημεία. Αναφερόμαστε στην ανάγκη δημοκρατία δημοκρατικών δικαιωμάτων, αποφυγή διάκρισης, προώθηση ποικιλομορφίας, της διαφορετικότητας και να λάβουμε υπόψη και την απειλή του Brexit στα πλαίσια των, ε, της Βορείου Ιρλανδίας και των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στη Βρετανία. Θέλαμε να φέρουμε βασικά στοιχεία λοιπόν. Ίσως λόγω του ορίου ε, του κειμένου να έχουμε κάποιες παραλήψεις μπορούμε να το συζητήσουμε και να επεκταθούμε μέσω τροπολογιών. Παρακαλώ τους ευρωβουλευτές να συνεργαστούν ούτω ώστε να καλύψουμε όπως το αρμόζει το θέμα της ηθαγένειας και να προστατεύσουμε τους πολίτες. Όπως είπατε και στην αρχή, στην εισαγωγή, θέλουμε οι πολίτες να είστε επίκεντρο της προσπάθειας. Θέλω να υπενθυμίσω στα μέλη και του Κιώδη ότι οι τροπολογίε μέχρι Τετάρτη 14 του μηνό πρέπει να υποβληθούν. Χάσαμε κάποιε προθεσμίε, αλλά προσπαθούμε να τηρήσουμε την προθεσμία του Δεκεμβρίου για να ψηφίσουμε, ίσω ούτω ώστε στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου να υποβληθεί το θέμα. Οι τροπολογίε και όλη η διαδικασία ίσω να είναι περιορισμένα χρονικά. Θα συνεργαστούμε στην Γραμματεία να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν φταίμε εμεί που ακυρώθηκε η συνάντηση προηγούμενη. Γι' αυτό καθυστερήσαμε. Και γι' αυτό έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Ευχαριστώ, Ματίνα. Κάποιοι σκιώδεις είναι παρόντες. Κύριε Βίστεσεν από το ECR, θέλετε να πείτε κάτι. Από πλευράς ECR είναι ξεκάθαρο. Η Θαγέννη Σοπρακής Ενώσεως συμπληρώνει την εθνική θαγένεια. Μόνο αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν να δώσουμε κάποια δικαιώματα στην ευρωπαϊκή θαγένεια με τον τρόπο που προσεγγίζεται. Το εκλογικό νόμος είναι εθνική αρμοδιότητα και έτσι πρέπει να παραμείνει. Και όσον αφορά και τι ευρωεκλογέ, θα υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίε. και θα προσπαθήσουμε μαζί με την εισηγήτρια να καταλήξουμε σε συμβιβασμό επ' αυτού. Άλλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, όχι, όχι. Ίσως ένα σχόλιο, κάτι της Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατη. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Υπενθύμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη θητεία της έχει εκδώσει σχετική έκθεση για την Ιθαγένεια και έκθεση για την πρόοδο για τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Υπήρξε και έκθεση σχετική του Κοινοβουλίου όσον αφορά το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και και τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη θητεία τη για να προωθήσουμε τα δικαιώματα τη ευρωπαϊκή ηθαγένεια, κυρίω τα εκλογικά δικαιώματα. Εκεί βάλαμε δέσμη μέτρων και προτάσεων το Δεκέμβριο για την ελεύθερη εξαγωγή των εκλογών στην Ένωση, κατά τα λοιπά για το σεβασμό των δικαιωμάτων ατόμων που ανήκουν σε μειονότητε, βασικό βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που είναι στη χάρτα και στη συνθήκη. Εμείς δεν έχουμε γενικές εξουσίες για τις μειονότητες. Δεν δίνω λεπτομέρειες, αλλά μπορώ να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Εκλογικά θέματα. Αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών γενικά. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και υπάρχει νομολογία του ΔΕΚ. Όπως η υπόθεση Τελβίν για τον ορισμό τη σύνθεση του εκλογικού σώματος αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι αυτή. Σύμφωνα με την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, κυρίω με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οπότε, η ε, ψηφοφορία από ε, εξαποστάσεως. Το Κοινοβούλιο ήθελε να αναδιαμορφωθεί ο σχετικό εκλογικό νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το σημείο δεν θεωρείται ότι δημιουργεί νομική υποχρέωση αυτά και με τα χαράς να απαντήσω. Σα ευχαριστώ πολύ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο προορισμό για την έκταση των χρηματοδοτήσεων, νομίζω ότι καλό θα είναι να διευκρινίσουμε τι είναι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια και τι σημαίνουν όλα αυτά τα δικαιώματα δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να κάνετε κάποια καταλητικά σχόλια. Ναι, κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι πιο πολλοί, αν όχι όλοι οι συνάδελφοι, θα συμφωνήσουν ότι το Brexit και η άνοδο τη ακροδεξιά ε, αποτελούν μια πραγματική απειλή για την έννοια της ε, ηθαγένειας. Γι' αυτό πιστεύω ότι η γνωμοδότηση και το θέμα αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, πιο έντονη από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Και παρά τις περιορισμούς, θα σας σύστηνα στην άδελφη να συμμετέχετε στην διαδικασία αυτή και έχω υπόψη μου ότι πλησιάζουν οι εκλογές, ε, αλλά έχουμε και 22 κρατημέλη τα οποία δεν περιορίζουν από τους πολίτες του το δικαίωμα της ψήφου όταν ε, μένουν σε άλλο κράτος μέλος. Ε. Αλλά έχουμε και τέτοια κρατημέλη που περιορίζουν αυτό το δικαίωμα του ψηφίζουν στα, στους πολίτες που μένουν σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό προφανώς αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αλλά δεδομένη τη ανόδου τη ακροδεξιά, νομίζω ότι καλό είναι να τονίσουμε με σωστό τρόπο τη σημασία του θέματο αυτού στην τρέχουσα χρονική στιγμή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Σεσίλη, θέλεις να πάρεις το λόγο γιατί ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Αν συμφωνείς Μαρτίνα να ακούσουμε την κυρία Κίνγκε. Σεσίλ για τη γνωμοδότηση για την υπηκότητα. Στο θέμα της κυρίας Άντερσον, λοιπόν. Είσαι σκιώδης από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ ε, την κυρία Άντερσον για το σχέδιο γνωμοδοτήσεώς της. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια πράγματι είναι νομική πραγματικότητα που ενισχύει και προωθεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα, εμπλέκοντας τους πολίτες στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Εκτιμώ την αφορά που κάνει η συγκίτρια στο άρθρο 2 της Συνθήκης Ένωσης και στα άρθρα 21 και 22 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Να προσθέσω σχετικά με αυτό και ότι σε μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι αλλοδαπείς αλλοδαποί πολίτες Ένωσης με άδεια διαμονή ε, μακρά διαρκεία ε, μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Θα πρέπει να προστατεύει τι μειονότητε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι πολίτε τη Ένωση έχουν δικαίωμα ψήφου στο, όσον αφορά το Ευρωκοινοβούλιο και οι χώρε που δεν σέβονται αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κυρώσει. Η διαφορά ετικότητα είναι αδιαφεσβήτη αξία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είναι αρχή που θα πρέπει να τύχει εγγύσεων, όχι μόνο μέσω των εκλογών, αλλά και μέσω των πολιτικών ένταξης. Και γι' αυτό προσέθεσα μια υπενθύμηση στην οδηγία που εξισώνει τους πολίτες με άδεια διαμονής μακράς διαρκείας με την κατάσταση Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να, να προστατευθούν ε, οι πολίτες από γλωσσική διάκριση, αλλά πολλές άλλες μορφές διάκρισης πρέπει να καταπολεμηθούν ε, εξίσου θα παρουσιάσω σχετικές τροπολογίες. Έτσι να εγγυηθούμε τα δικαιώματα όλων, δηλαδή να είναι πλήρης η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να προστατεύει όλους τους πολίτες. Πολίτες, όπως προανέφερα, με άδεια διαμονής μακράς διαρκείας, θα πρέπει και αυτοί να επισέλθουν σε αυτήν την τροποποίηση του κανονισμού, σε πλήρη σεβασμό του άρθρου 2 uh, ε, της συνθήκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σεσίλ. Και τώρα η Τζιν. Μια και καταφτάσατε. Αυτή η γνωμοδότηση η αίσθηση έχει κάνει. Όλοι μπαίνουν σιγά σιγά στο προσκήνιο. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κυρία Λάμπερτ ε, από τους πράσινους. Είστε σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα για το θέμα αυτό. Και ναι, προφανώς καλώς ορίζουμε τη γνωμοδότηση της ε, Μαρτίνα Άντερσον και εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε η κυρία Κιέγγε για το πώς αυτό ισχύει και εφαρμόζεται στα άτομα με δικαιώματα μακράς παραμονής. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα θέλαμε να προσθέσουμε. Ένα από αυτά είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει σιγά σιγά προσοχή στο τι συμβαίνει στα παιδιά των οποίων οι γονείς ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπει η συνθήκη, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο να καθερθεί το δικαίωμα, να καταχρηθεί το δικαίωμα ψήφου στις χώρες που μένουν και σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και πιο αυστηροί οι κανόνες για την ηθαγένεια. Είναι λοιπόν δύσκολο να γίνουν όλα αυτά αν ζει κανείς εκτός της χώρας ε, της εθνικότητάς του λόγω του επαγγέλματος των γονιών του. Να το έχουμε υπόψη μας τουλάχιστον. Το δικαίωμα επίση για την οικογενειακή ζωή για άτομα με ηθαγένεια ευρωπαϊκή Ένωση που βρισκόνται σε σταθερή σχέση είναι παντρεμένα με άτομα εκτό Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι ανεπαρκη και ελλειπη η εφαρμογή αυτού. Και αυτό λοιπόν έχει να κάνει με τα ταξίδια εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Να επιστήσω επίση την προσοχή στη ανάγκη να υπάρχει αναλογικότητα από πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι απαφώσει για την ε, αφαίρεση ε, και την ε, επιστροφή ατόμων χωρίς ηθαγένεια. Και εδώ χρησιμοποιείται πολύ συχνά το τεκμήριο των άστεγον, ότι κάποιο είναι άστεγο και βλέπουμε ότι υπάρχουν και σχετικέ αποφάσει του δικαστηρίου και θα ήθελα λοιπόν να τα πάρουμε υπόψη αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και ο Πρόεδρο. Ήταν ε, πολλέ ε, οι παρατηρήσει σα και πλούσιο το περιεχόμενο αυτών σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Προφανώ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα ποτέ Και δεν ξέρω πώ θα τα βάλουμε όλα αυτά σε μια γραμματότηση. Αλλά φυσικά η γνωμοτότηση θα πω, Σε εφαλτήριο για μια γενικότερη συζήτηση. Ωραία. Άννα, τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Πώ λαμβάνεται υπόψη τα όσα έχει ανακαλύψει για τις ε, χρυσές ε, θεωρήσεις και της ε, χρήσης ε, της έννοιας της ευρωπαϊκής υπηκότητας για σκοπούς ε, πέρα από το ξέπλυμα χρήματος ε, για οικονομικούς σκοπούς, νόμιμους και μη. Χτες στο Μονακό έγινε μια σύλληψη, πληροφορήθηκα, ενός Ρώσου πολιτή Ριμπόλοβλεφ, ο οποίος είχε πάρει κυπριακή υπηκότητα το 2012, η γυναίκα του δε και η κόρη του είχαν διάφορες υπηκότητες και ασφαλώς πρόκειται για έναν κυρίο με πολλά χρήματα, με ποδοσφαιρική ομάδα που θα μπορούσε να υποστηρίζει την προεκλογική εκστρατεία όπως ο Άρεν Μπάνκ στην ε, Βρετανία υποστήριξε το Brexit και έτσι με τον τρόπο αυτό παρεμβαίνει και επεμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική και Στι ευρωπαϊκέ εκλογέ στην επιλογή του Ευρωπαίου πολίτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν το λαμβάνει υπόψη αυτό. Λαμβάνει υπόψη τέτοιου είδου απειλέ. Μάλιστα λέει ο πρόεδρο, ε, δημιουργικότατη παρέμβαση. Σχόλια εκτό μικροφώνου, η κυρία Γκόμες. Μάλιστα, χρυσέ ε, βίζες, χρυσέ θεωρήσει, λέει ο πρόεδρο. Δεν ξέρω. Κατά κάποιο τρόπο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή. Αλλά. Δεν ξέρω. Θέλετε να απαντήσετε, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ε, όχι, εσεί η ίδια. Πείτε μας κάτι για αυτές τις ε, Golden Visas. Ε, ευχαριστώ. Και δεν θα μπω σε μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας, αλλά να πω ότι υπάρχει και η έκθεση για την Ιθαγένεια, την παρουσίαση Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι και λαμβάνει υπόψη τι δεσμεύση να αξιολογηθεί η ευρωπαϊκή θαγένεια και οι αξίες αυτής και να περιγραφεί τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, να περιγραφεί οι ευρωπαϊκές, να περιγραφούν οι ευρωπαϊκές και οι πρακτικές και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και συγγνώμη, ο σκοπό τη Ευρωπαϊκή και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δημοσιευτεί αυτή η έκθεση πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα, ωραία μα τράτε και τα καταλαβαίνουμε, λέει ο πρόεδρο. Πολύ καλά. Η προθεσμία για τα κατάσταση οπολογιών είναι τροπολογιών είναι η 14 Νοεμβρίου και είναι σαφές ε, πόσο επίκαιρη είναι αυτή η γνωμοδότηση και πόσο ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους κοιόδες. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Συνεχίζουμε. Είμαστε στην ώρα μας. Είναι εδώ και ο κύριος Ουγγουρεάνου. Έχουμε την παρουσίαση από την Επιτροπή δύο προτάσεων σχετικά με σύναψη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχίας διαμονής για τους κατόχους κοινών ε, διαβατηρίων και για τους κατόχους διπλωματικών υπηρεσιακών και επίσημων διαβατηρίων. Παρακαλώ. Ναι, Όντω, πρόκειται για το θέμα που είπατε, σύναψη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Βραζιλία ε, για υποχρέωση θεώρηση βραχία διαμονή ε, για του κατόχου διαβατηρίων. Η μία και η άλλη μου έκθεση έχει να κάνει για του κατόχου διπλωματικών υπηρεσιακών και επίσημων διαβατηρίων. Πρόκειται για τον ε, κανονισμό 601, ο οποίο εισάγει κάποιε αλλαγέ στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάει για διάρκεια επιτρεπόμενης διαμονής 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περίοδο 180 ημερών. Είναι αναγκαίο λοιπόν τέτοιες συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βραζιλία να συμπεριλαμβάνουν τους νέους ορισμούς. Για να υλοποιηθούν λοιπόν αυτοί οι νέοι ορισμοί όσον αφορά τη βραχία διαμονή, τον Ιούλιο του 2014 ενέκρινε σύσταση Επιτροπή για απόφαση του Συμβουλίου προκειμένου να ανοίξουν ε, διαπραγματεύσεις για να τροποποιηθεί η συμφωνία αυτή όσον αφορά την υποχρέωση θεώρηση βραχίας διαμονής και το Συμβούλιο την ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2014. Μετά λοιπόν την έγκριση από το Συμβούλιο ξεκίνησε διαπραγματεύσεις η Επιτροπή για να τροποποιηθεί αυτή η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης και τον Οκτώβριο του 2014 εγκρίθηκε, ε, κατέληξε η διαπραγμάτευση. Τώρα βεβαίως η εισηγητής εννοείται ότι συστήνω τη σύμφωνη γνώμη. Η παρουσίαση του σχεδίου μου στην Επιτροπή θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Δεκεμβρίου και κατά πάσα πιθανότητα 10 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε κύριε Γκουριάνου. Υπάρχει καμία αντίδραση, δεν κάτι να πείτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγα έχω να προσθέσω. Απλώς θέλω να επενθυμίσω ότι υπάρχουν όντως δύο διαφορετικές συμφωνίες που ισχύουν όσον, ε, αφορώ, όσον αφορά την ε, εξαίρεση αυτή, την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης βραχίας διαμονής και ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν από την λήξη της θητείας αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να έχει τροποποιηθεί ορισμός οριστικά και αντί να ισχύει τρει μήνες μέσα σε έξι μήνες, να είναι αυτή η βραχία διαμονή, να αλλάξει και να γίνει αυτό που είπαμε, δηλαδή 90 μέρες μέσα σε ένα διάστημα 180 ημερών. Αυτές οι δύο συμφωνίες με τη Βραζιλία πάντως ακολουθούν την ίδια ακριβώ προσέγγιση όπως άλλες έξι τροποποιημένες συμφωνίες που έχει εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επίσης τροποποιούν την ε, διάρκεια της βραχής διαμονής που εκτελεί την Παχάμας, Σεχέλες, Μαυρίκαιος και άλλες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για έξι τέτοιες συμφωνίες. Την ίδια ακριβώ προσέγγιση ακολουθεί και η τροποποίηση τη συμφωνία με τη Βραζιλία. Πήρε περισσότερο χρόνο να έρθει στο Κοινοβούλιο εξαιτία καθυστερήσεων από πλευρά τη Βραζιλία. Και επίση να πω ότι αυτέ οι ποιημένες ε, συμφωνίες θα αρχίσουν να ισχύουν άπαξ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του και έχουν κυρωθεί και από τη Βραζιλία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Θέλεις να πεις κάτι. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει κυρία Βεζιά. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Πρόκειται για τεχνικές ε, διευθετήσεις και επιτέλους για μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόλαβε πριν αρχίσει να ισχύουν αυτές οι συμφωνίες συστηματικά, αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Αλλά δυστυχώ δεν συμβαίνει συστηματικά. Οπότε για μια φορά που τα πράγματα είναι όπως πρέπει, α το υπογραμμίσουμε. Ας πούμε και τα καλά. Ευχαριστούμε, Κριστίν, που είσαι και εσύ σκιώδης για αυτό το θέμα. Άννα, τι έχεις να πεις. Δεν έχω αντίρρηση για τη Βραζιλία. Αντίθετα, πιστεύω ότι όντως πρέπει να διευκολύνουμε τους Βραζιλιάνους να ταξιδεύουν στην Ευρώπη και ελπίζω ότι και η χώρα μου θα τους διευκολύνει ακόμα περισσότερο για να έρχονται σε μας. Ζούνε δύσκολους καιρούς στη χώρα τους με τον νέο πρόεδρο. Αλλά η ερώτησή μου πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις άλλες συμφωνίες που είπατε ότι με αυτές συμφώνησε το Κοινοβούλιο πρόσφατα. Όλες αυτές όμως τις δικαιοδοσίες τις έβαλε όσα ε, πρόσφατα σε μια μαύρη λίστα. Ακριβώς για το θέμα των χρυσών θεωρήσεων. Και την αγορά της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Αυτό το λαμβάνει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της το λαμβάνει υπόψη πριν ζητήσει από το Κοινοβούλιο τη σύμφωνη γνώμη. Αλλιώς νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να λάβει υπόψη του αυτή τη διάσταση του ζητήματος. Πρόεδρος. Ωραία. Ένα τελικό σχόλιο, αν θέλει, ο εισηγητής όχι. Εντάξει. Οπότε τελειώνουμε με αυτό το σημείο και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε για τα σχόλιά σας και για το έργο σας. Οπότε συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στο Α, είναι εδώ κυρία Κινίτσι, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με το σημείο 7 που είναι η παρουσίαση σχεδίου έκθεσης για πρόταση που έχει να κάνει με το άσυλο και το αμύφ. Υπάρχουν τροπολογίες ε, για τον κανονισμό άμυφ, προκειμένου οι χώρες μέλη να μπορούν να χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα κονδύλια για να αντιμετωπίσουν τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης η πρόταση επιτρέπει στις μέλη να δεσμεύσουν ποσά στα δικά τους εθνικά προγράμματα αναθεωρώντας ε, τα. Οι συντονιστέ συμφώνησαν να δουλέψουν πάνω σε αυτή την πρόταση μόνο στα αγγλικά γιατί η διαδικασία δεν προβλέπει πολύ χρόνο για να μπορέσει πριν τα τέλη της χρονιάς να εγκριθεί αυτή η πρόταση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Κινίτσι, η οποία αντικαθιστά την ε, εισηγήτρια και θα μας παρουσιάσετε κύρια στοιχεία του σχεδίου αυτού έκθεσης. Ευχαριστώ Καταρίνα και έχεις και το λόγο. Ευχαριστώ Κλοντ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπε και ο Κλοντ, με τον λόγο εν ονόματι της Νταλή, που είναι η συγγήτρια όσον αφορά για την χρήση αυτών των ποσών για τον τομέα της προστασίας ε, να βοηθήσουν την Ιταλία και την Ελλάδα για το θέμα της μετανάστευση. Ζητεί συγγνώμη κυρία Νταλή, από όλους τους που απουσιάζει σήμερα και δεν παρουσιάζει την έκθεση. Δυστυχώ όμω είχε ανηλυμένε υποχρεώσει. και δεν κατάφερε να αποδεσμευτεί. Ο κανονισμό τροποποιεί το Ταμείο για το Άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη και το άρθρο 18 του κανονισμού. Η κυρία Μυριαμνταλή εξηγεί ότι μετά τη μετασταυτική κρίση του 2015, 843 εκατομμύρια ευρώ από πλευρά του ΑΜΙΦ δεσμεύτηκαν για την μετεγκατάσταση ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασία από την Ελλάδα και την Ιταλία και για την ένταξη των Σύρων και να έρθουν και οι Σύροι πρόσφυγες στην Τουρκία. Τα 843 εκατομμύρια ευρώ που δεσμεύτηκαν για το 2016 για εθνικά προγράμματα των κρατών μελών στα πλαίσια του ΑΜΙΦ παραμένουν διαθέσιμα από αυτά πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ το 843. Σύμφωνα με τους κανόνες, οι πληρωμές θα έπρεπε να δοθούν μέχρι το τέλος του 2018 για τους στόχους που είχαν τεθεί. Μετά από αυτό η χρηματοδότηση δεν θα είναι διαθέσιμη για τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των εθνικών προγραμμάτων του ΑΜΙΦ. Για να εγγυηθούμε ότι οι πόροι που δεν χρησιμοποιήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων του ΑΜΙΦ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τεχνικές τροποποίησεις του άρθρου 18 του κανονισμού. Στο σχέδιο εκθέσεω, η κυρία Μίρια Μνταλή δίνει 20% ελάχιστο για τη μεταφορά των ετούντων διεθνούς ασύλου και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Η συγγήτρια θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη που προτίθενται να συνεχίσουν να μεταγκαθιστούν άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας δεν θα πρέπει να αποθαρρυνθούν. Κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το Συμβούλιο αρχικά προέβλεπε υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν 160.000 ανθρώπους από την Ιταλία και την Ελλάδα. Άλλε αποφάσει μείωσαν τη μεταφορά περίπου σε 98.000 ανθρώπου. Οι αριθμοί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν ότι πόρα απέχουμε από την επίτευξη των αλόγων αριθμών. Αυτό σημαίνει ότι πολλά απομένουν να γίνουν και τα κράτη-μέλη που θέλουν να συνεχίσουν ή να επενδύσουν περισσότερα στη μετεγκατάσταση ε, δεν θα πρέπει να βρεθούν σε δυσμενή θέση. Πιστεύει η ότι οι απομένοντες πόροι θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε δράσεις και μέτρα που αντικατοπτρίζουν την αρχή της αλληλεγγύης ε, και του διαμοιρασμού των ευθυνών ε, για τα κράτη-μέλη. Πάνω σε αυτό η κυρία Μίρια Μνταλή προτείνει να αναφέρονται ποσοστά που θα εγγυηθούν ότι τουλάχιστον το 20% των ποσών που πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν θα δοθούν για την ενίσχυση και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού κοινού συστήματος ασύλου. Και άλλο 20% για την υποστήριξη της νόμιμης μετανάστευσης και να προωθηθεί και η κατάλληλη ένταξη των πολιτών που μεταναστεύουν από τέτοιες χώρες. Θέλει να υπογραμμίσει η κυρία Νταλή ότι θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν οι διθεσμοί πόροι, αλλά αρχικό στόχο τη μετεγκατάσταση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει ξεχωριστά και να παραμεληθεί. Τα κράτη-μέλη που σεβάστηκαν τι ποσοστώσει μετεγκατάσταση δεν θα πρέπει να βρεθούν σε δυσμενή θέση μέσω των δράσεων των κρατών μελών. Η κυρία Νταλή θέλει να συνεργαστεί με του και σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε αυτή η έκθεση μέχρι τέλου του έτου να είναι έτοιμη. Έτσι θα εξασφαλίσουμε την ανακατανομή των πόρων για τους ε, κοινά υποστηριζόμενους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατρίνα, ευχαριστώ που αντικαθιστά την κυρία Ντάλη για το σημαντικό αυτό θέμα. Από τους Κιώδης που είναι εδώ. Είναι κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο. Κριστίν, Κριστίν Βεργιά, θέλεις να λάβεις το λόγο. Εκ μέρους της κυρίας θα μιλήσω. Ορίστε, λέει ο πρόεδρος. Η συνάδελφος Μαρίν Μπιόρκ ζητά συγγνώμη που απουσιάζει. Μου στη το κείμενο της παρέμβασής της. Να διαβάσω. Να ευχαριστήσω την συγγήτρια Μίρα Μταλή για την έκθεσή της που μας διβιβάστη γνωρίζουμε την πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή η διαδικασία. Και σε αυτό το πλαίσιο η συγγήτρια προτείνει τις σχετικές τροπολογίες. Το χαρτοφυλάκιο δεν τεχνικής φύσης, όπως το παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχής, γιατί μένουν 507 εκατομμύρια ευρώ από τα 843 εκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί για τη μετακατάσταση των ετούντων άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα. Το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του 2017 με τον τίτλο να επιτρέψουμε τη μετακατάσταση έκανε τα εξή αιτήματα και αν αυτά είχαν ληφθεί εισακουστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχαμε την παρούσα κατάσταση. Το Κοινοβούλιο ζήτησε δύο στοιχεία βασικά. Μεταγκατάσταση από Ελλάδα όλων των επιλεξίμων που κατέφτασαν μετά τις 20 Μαρτίου του 2016, κάτι που δεν έγινε παραβιάζοντας την απόφαση μετεγκατάστασης. Η παράταση των μέτρων μετεγκαταστάσεως μέχρι την έγκριση της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου. Ήταν κάτι που ζητήσαμε. Βασικό στοιχείο να ζητήσουμε επέκταση της ομάδας των επιλεξίμων ανθρώπων όπως του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς όμως έγινε αυτό πολύ, πολύ αργά στη νέα πρόταση. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσέθεσε στους δικαιούχους της νέας προτάσεως εκείνους που χρήζουν διεθνή προστασία. Αν τα κριτήρια επιλεξιμότητας είχαν εφαρμοστεί από το 2015 θα είχαμε αποφύγει την παρούσα κατάσταση που είναι καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα όπου δύο ομάδε ετών τον άσυλο έχουν εξαιρεθεί από το μηχανισμό. Η ΠΚΟΗ e από το Αφγανιστάν και το Ιράν χωρί να αναφέρουμε τον αποκρισμό πολλών ανθρώπων σε κατάσταση εξαιρετικά ευάλωτη, ανεξάρτητη εθνικότητα μεταξύ αυτών πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι. Λοιπόν, εφαρμόζοντα το μηχανισμό ελληνική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γίνει αυτό πρέπει να συνεχιστεί η λειτουργία του μηχανισμού μετεκαταστάσεως των ετούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Πιο σημαντικό αυτό. Γι' αυτό, μέσω των σχετικών τροπολογιών, ζητούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα ποσά να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μόνο από τα κράτη-μέλη εκείνα που θέλουν να μεταγκαταστήσουν δικαιούχους ασύλου και όχι μόνο την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες όπως είναι η Ισπανία ή Μάλτα αυτοί οι πόροι εγκρίθηκαν για ένα μόνο στόχο, για αλληλεγγύη. Δεν είναι αποδεκτό για μας να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς καταστολής όπως η καταναγκαστική επιστροφή, ο αναπατρισμός. Ευχαριστώ πολύ, Κριστίν. Και να ακούσουμε τι μας λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα. Συγγνώμη, γιατί έφτασα τρέχοντα. Έχω λαχανιάσει. Σα ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και για το σχέδιο τη έκθεση, το οποίο ασφαλώ ε, το καλωσορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σα υπενθυμίσω ποιο έχει η τρέχουσα ε, κατάσταση, το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο για την επανεκατάσταση. Ξέρετε ότι έχουν ε, πάρει τέλο ε, οι σχετικέ αποφάσει για επανεκατάσταση. Δεν υπάρχει λοιπόν οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο για υποχρεωτικέ τέτοιε επανεκαταστάσει. Προφανώ όμω το συζητάτε αυτό και εξετάζετε το θέμα αυτό, αλλά δεν έχει συμφωνηθεί κάτι επίσημα ακόμη. Και έτσι. Δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις που συνολικά. Και έτσι λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει κάτι πολύ ε, υποφελές. Να συνεχίσει η υποστήριξη της ε, θελούσιας επανεκατάστασης. Είναι σαφές ότι η πρόταση αυτή ε, κινείται προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αλληλεγγύης και ξέρουμε και ότι λήψη νομοθετικού πλαίσιου για το θέμα αυτό, ο αριθμός των ε, επανεκαταστάσεων δεν θα είναι υψηλός. Θα είναι μάλλον περιορισμένος. Και ως εκ τούτου γνωρίζουμε ότι θα είναι επίσης πολύ σημαντικό τα κονδύλια αυτά να χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, να μπορούν να χρησιμοποιούνται δηλαδή και για, άλλα, άλλους σκοπούς, όπου ενδεχομένω να είναι πολύ προφανής και επίγουσες οι ανάγκες, όπως για παράδειγμα άσυλο, ενσωμάτωση, οποιαδήποτε επένδυση σε άσυλο και ενσωμάτωση είναι έκφραση αλληλεγγύης, αλληλεγγύης προς τους αντούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και προς τα κρατημέλη και στους διάφορες σχετικές ε, χώρες. Ε, οποιαδήποτε λοιπόν ε, επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή είναι ένδειξη εγγυλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα σε ό,τι αφορά την έκθεση ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να υποβάλει ετήσια έκθεση προς το Κοινοβούλιο για τη χρήση των πόρων αυτών. Είναι πάρα πολύ ε, θετική θεωρούμε αυτή η πρόταση στην έκθεση. Επίσης και τις άλλες προσθήκες ε, στις ιδεολογικές σκέψεις ε, που διευκρινίζουν, θεωρώ, τις διατάξεις αυτή η οκταετή περίοδος για έλεγχο από τις εθνικές βουλές. Αυτό το υποστηρίζουμε. Αυτό που δεν υποστηρίζουμε τώρα είναι η πρόταση για αλλάξει το ποσοστό μετακατάστασης, γιατί αυτό τι θα σημαίνει. Ότι χρησιμοποιούμε ουσιαστικά το άμεφ για να αντικαταστήσουμε τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου. Αν θέλουμε μια αντιστοιχεία για μια υποχρεωτική ποσόστοση επανεγκατάστασης. Ξέρουμε βέβαια ότι αυτό δεν θα γίνει δεκτό, γιατί τέτοιες συζητήσει έχουν γίνει και δεν έχει υπάρξει ακόμα λύση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Δουβλίνου. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε η πρόταση αυτή να καταστεί και βιώσιμη. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα ποσοστά αυτά δεν είναι άκαμπτα Άρα, αυτό θέλουμε να κάνουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσουμε την, ε, από την Επιτροπή σα να φροντίσει η πρόταση αυτή να γίνει αποδεκτή για να εγκριθεί μέχρι το τέλη του έτους. Και έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι πάρα πολύ αντεπορογωγική η πρόταση για ελαχιστά ποσοστά επανεγκατάστασης. Και κατά τα άλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προτάσεις σας και αν έχετε ερωτήσεις, με χαρά να τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ναι, έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω, μήπως η κυρία Κινίτσι έχει ερωτήσεις. Ή θα απαντήσετε τώρα ή θα περιμένουμε όταν έχουμε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ όπως αναφέρθηκε, δεν τεχνικής φύσεως, αλλά πολύ ευαίσθητο και περίπλοκο χαρτοφυλάκιο. Άρα καλό θα ήταν να είναι η συνάδελφος Μίρια Μνταλή παρούσα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε, ε, εκείνη πρέπει να αντιδράσει στις συνεισφορές και τις απόψεις για να μπορέσει να συνεχίσει την εργασία της. Ευχαριστώ. Okay, Ωραία, είναι εδώ η βοηθή της, θα τα σημειώσουν όλα αυτά. Μαρή Κριστίν, θέλεις να απαντήσεις. Έχω μια μικρή διευκρίνηση που θέλω. Γιατί δεν καταλαβαίνω τόσο καλά τη θέση της Επιτροπής. Αν κατάλαβα καλά, αλλά επειδή δεν είμαι επίσημα σκιώδης, μπορεί και να ασφάλω. Αν κατάλαβα, οι τροπολογίες δεν προβλέπουν ποσοστώσεις, γιατί αυτό το κόκκινο πανί, από ό,τι κατάλαβα στη συζήτηση, και η συγγήτρια και οι σκιώδες κουνάνε όντως το κόκκινο πανί κάθε φορά, ενώ θέλουμε να προχωρήσουμε. Εμείς μιλάμε για αποθεματικό που είχε προβλεφθεί έτσι κι αλλιώς, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χώρες σε θελοντική βάση. Ήδη ισχύει. Το μόνο που ζητάμε είναι να υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση, κυρίως δεδομένης της εξέλιξης των μεταναστευτικών ρευμάτων. Ξέρουμε ότι δεν είναι πια μόνο Ελλάδα και Ιταλία, γιατί οι μετακινήσεις ε, μεταφέρονται, ακόμα και αν το μεταφέρονται δεν είναι σωστός όρος, και στην Ισπανία. Οπότε η απάντηση της Επιτροπής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των τροπολογιών, εκτός αν σφάλω κάπου. κύριε Κινίτσι. Και εγώ συμφωνώ με την απορία της συναδέλφου. Άκουσα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω απορίες, αλλά νομίζω η κυρία Μίρια Μνταλή θα επανέλθει και θα συνεργαστεί για να αποσαφινιστούν αυτά. Έτσι που παρουσιάστηκε το θέμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν φαίνεται να δόθηκαν απαντήσεις επί της ουσίας και για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Δεν μας εκάλυψε πλήρως η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά η κυρία Αντάλη θα μπορούσε να διευκρινίσει. Yeah. Καλώς. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα η συγγήτρια όντω να το ξεκαθαρίσει τα χρήματα που θα πηγαίνουν στη μετακατάσταση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. θα ήθελα αυτό να εμφανίζεται στις τροπολογίες. Το είπε και η Μαρή Κριστίν και εσύ Κατρίνα που αντικαθιστάς τώρα την εισηγήτρια. Αυτό θα πρέπει να το μεταφέρεις ξεκάθαρα στην εισηγήτρια και είμαι σίγουρος ότι θα δείξει κατανόηση. Και φυσικά πρέπει να το ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας ακούει, οπότε το ξέρει. Καλώς, Ευχαριστούμε και την Μαρή Κριστίν και εσένα, Καταρίνα. Τώρα, προθεσμία για την υποβολή τροπολιών είναι 12 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που αντικαταστήσατε την εισηγήτρια και έτσι μπορέσαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αυτό το σημείο. Τώρα έχουμε περίπου τελειώσει. άγγερα. Κάτι που δεν είναι εύκολο, πέμπτη πρωί. Ο κύριος Τερικάμπρας δεν είναι εδώ, γι' αυτό δεν ξέρω ή έρχεται, που είναι το τελευταίο μας σημείο. Γι' αυτό το τελευταίο σημείο, συνάδελφοι. Έρχεται ο κύριος Τερικάμπρας. Είναι στον δρόμο. Οπότε τι να κάνουμε. Θα σταματήσουμε, θα διακόψουμε για 20 λεπτά. 20 λεπτά ακριβώς διακοπή. Στις 10 και μισή να είσαστε πάλι εδώ για να ξεκινήσουμε με αυτό το τελευταίο σημείο. Okay, thank you. Thank you for your patience. Okay, thank you very much, colleagues, and thank you, Mr. Terry Cabras, um, for, um, for getting here and... it's μπορούμε να συνεχίσουμε. Όντω, 10 και 40 είχαμε προβλέψει το θέμα σα. Τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά πέμπτη πρωί. Πάμε καμιά φορά πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπουμε. Ευχαριστούμε πάντως που ήρθατε και ευχαριστώ όλους σας για την υπομονή σας. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το σημείο 8. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσία του σχεδίου γνωμοδότησης του κυρίου Τερικάμπρα όσον αφορά την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Είναι μια πρόταση που βασίζεται στο κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αξίες του και το γεγονός ότι όλα αυτά αποτελούν την βάση της ίδιας της ύπαρξης και του σεβασμού του κράτους δικαίου. Οπότε η Επιτροπή μας δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε πρόσφατα και των εξελίξεων όσο αφορά το κράτος δικαίου και την προστασία και την πρόθεση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε Τερικάμπρας. Παρακαλώ, παρουσιάστε μας το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας και ευχαριστώ πολύ και τους συναδέρφους. Αυτό το μέσο, το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, πρόκειται για μια καινοτομία όσον αφορά τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει να κάνει και με πέρα από την περίοδο μέχρι το 2020. Συνεπώς ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρότασή της με μέτρα υπέρ του κράτους δικαίου στις χώρες μέλη, ώστε να γίνονται σεβαστές οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγχρόνως όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται δεν θα πλήττουν απευθείας τους ε, πολίτες. Ευχαριστώ λοιπόν τους εισηγητές Μπάτς και Κόντ των ε, επί αρμοδίων επιτροπών δηλαδή και σας ε, πρόεδρε που ζητήσατε την παράταση της προθεσμίας γιατί η πρόταση αυτή πρέπει να εξεταστεί σε βάθος ακριβώς επειδή είναι καινοτόμα και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας. Τώρα όσον αφορά την ουσία της πρότασής μου. Για τα άρθρα 2 και 3 πιο συγκεκριμένα έχουμε επιμερισμένη αρμοδιότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα θέλαμε, αντί να μιλάμε για το κράτος δικαίου, εμείς προτείνουμε την οριζόντια αντιμετώπιση αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, επίσης, στον ορισμό των ε, αδυναμιών όσον αφορά τις αξίες της Ένωσης, εμείς θέλουμε την ε, εξή προσέγγιση. Σε μια κατάσταση όπου υπάρχει συστημική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άπαξε και οι αρχές της Ένωσης υπονομεύονται άμεσα ή έμεσα με συστημικό τρόπο, είτε εξαιτία των πρακτικών, των παραλήψεων, των μέτρων ή ε, έλλειψης δράσης από τις αρμόδιες αρχές ή επειδή υπάρχουν γενικές πρακτικές ελλείψεις, έλλειψη δράσης λοιπά των αρχών που υπονομεύουν ένα ή πολλά ε, μέρη ε, που συνθέτουν το κράτος δικαίου ή τις αξίες της Ένωσης. Αυτό προτείνουμε για να εξηγούμε τι σημαίνει γενική έλλειψη όσον αφορά το κράτος δικαίου. Έρχομαι τώρα στο άρθρο 3. Εδώ παρουσιάζουμε τρεις περιπτώσεις όταν πρέπει να λαμβάνονται δηλαδή κάποια μέτρα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου. Δεύτερον, το 1 τρίτο των χωρών μελών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής υποβάλλουν μια αιτιολογημένη γνώμη στο Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνο σοβαρής απειλής σε μια συγκεκριμένη χώρα μέλος απέναντι ε, των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η τρίτο, το 1 τρίτο του Κοινοβουλίου της Επιτροπής ε, προτείνουν αιτιολογημένη γνώμη Επίσης, βάσει του άρθρου 7, αλλά παράγραφος 2, και την υποβάλλουν στο Συμβούλιο, αναφερόμενοι σε συνεχείς και επίμονες παραβιάσεις ε, του κράτους δικαίου των αξιών τη Ένωση, έτσι όπως αναφέρονται στο άρθρο 2. Η προηγούμενη πρόταση μιλούσε για σοβαρή παραβίαση και τώρα μιλάμε και για επίμονες ε, παραβιάσεις, επανειλημμένες. Ε, μετά την αξιολόγηση, την αξιολόγηση λοιπόν αυτών των γενικευμένων λήψεων ή παραλήψεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα πάνελ με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και ελπίζω να έχουμε τη βοήθεια και τη στήριξη των συναδέρφων για να βελτιωθεί αυτό το κείμενο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάμπρας. Είναι όντως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό και μια γνωμοδότηση για κάτι επίκαιρο και σημαντικό. Έχουμε το άρθρο 54 θα υπάρξουν λοιπόν συναντήσεις και δόνηση γειτών ε, στη συνέχεια. Ε, από το ΕΛΚ ο Σκιώδης μου έδωσε το εξή, αλλά προηγουμένως θα ακούσουμε τους υπόλοιπους Σκιώδης και μετά θα σας διαβάσω αυτό που μου έδωσε ο Σκιώδης της ΕΛΚ. Ε, Σεσίλ, παρακαλώ, από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης που προορισμό έχει την Επιτροπή Προπολογισμών και Ελέγχου Προπολογισμού. Έγινε πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή και σχετικά με την ομάδα μου πρέπει να πω ότι συμμεριστήκαμε μαζί του τη σημασία των αξιών που αποτελούν την ίδια τη βάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο σεβασμός των ελόγου αξιών πρέπει να είναι κάτι εγγυημένο σε όλες τις πολιτικές της Ενώσεως, συμπεριλαμβανομένου και του προπολογισμού αυτής. Στα πλαίσια αυτού ο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι προαπαιτούμενο, βασικό, για χρηματοπιστωτική, οικονομική, υγιή διαχείριση των οικονομικών και να είναι αποτελεσματική διαχείριση των δημοσιονομικών. Η πρόταση του εισηγητού είναι για νέα, αντικαθιστά το καθεστώ του δικαίου με αξίε τη ε, ενώσεω. Όσον αφορά τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια, συμπραγματεύονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτο δικαίου. Λοιπόν, οι γενικές ελλείψεις ε, αναφέρονται σε όλες αυτές τις καταστάσεις όπου υπάρχουν κίνδυνοι. Βρίσκω ενδιαφέρουσα την διαδικασία προβλέπου συγητής για την αξιολόγηση του καθεστώτος ελλείψεων της Ένωσης, όπως ε, και τα πάνελ για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Έδωσε απαντήσει ο συγητής και αυτές είναι σίγουρα ενδιαφέρουσες θα παρουσιάσω εν ονόματι τη ομάδας ε, των σοσιαλιστών τροπολογίες που θα έχουν στόχο να παγιώσουν τη θέση του, να ισχυροποιήσουν τη θέση του. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σεσίλ, ο κύριος Ντιούρεκ για το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν ε, θέλω να αναφέρω ότι τα άτομα αυτά ε, πρόκειται για περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ε, διαπίστωση της υπετιότητας. Σε μία πολιτισμένη λοιπόν κοινωνία υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας ως το σημείο που θα αποδειχθεί η ενοχή κάποιου ανθρώπου. Τίθεται λοιπόν το θέμα αυτό και αυτό είναι το θέμα όταν ασκείται πολιτική για την οποία δεν υπάρχει α, δημοκρατική εντολή. Οι κοινέ λοιπόν αυτές αξίες αναφέρονται στη συνθήκη. Είναι κοινέ αυτές οι υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα συζητάμε το θέμα αυτό για τις παραβιάσεις ε, από τις χώρες αυτές που κατηγορούνται για έλλειψη δημοκρατικού καθεστώτος και κράτους δικαίου, μία μέρα μετά από τις διαδηλώσεις και από τις δηλώσεις του κυρίου Φερχόφστατ κατά της Ουγγαρίας. Αυτή η εκστρατεία θεωρώ ότι προσβάλλει τους απογόνους της γενιάς του 56, προσβάλλει τις δημοκρατικές αξίες. Τέτοιοι πολιτική λοιπόν όπως ο κύριος Φερχόφστον θα πρέπει να τους υπενθυμίζουμε διαρκώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τσιφλική τους, είναι ένωση των κρατών μας. Δεν είναι πεδίο για τις ιδεολογίες του καθενός. και ο τρόπος ε, που λειτουργεί ουσιαστικά δικαιολογεί αυτά που βγαίνει και δηλώνει ο Ορμπάν για την, τις εποχές έλλειψης δημοκρατίας. Αυτή η μεταφιλελεύθερη λοιπόν τάση προκύπτει από την απόπειρα διαμόρφωσης του προϋπολογισμού και ε, λυπούμαστε και για τις δηλώσεις της κυρίας Ιντφέλντ για την Ουγγαρία. Κατηγόρησε την Επιτροπή Μπαρόσο για την υπερβολική προσήλωση της σε νομικίστικες διατάξεις και θα ήθελα, είπε, να είναι λιγότερο νομικίστικη η νέη, νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέτοια συζήτηματα συζητάμε λοιπόν σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. τέτοιες ιδέες δημοσιονομικών κυρώσεων θα πρέπει να καταργηθούν το συντομότερο δυνατόν. Σκιώδης τώρα για την ΚΟΕ είναι η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον Τέρι Κάμπρας, για τη δουλειά του και για την παρουσίαση. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εν πρώτης, να σταθώ σύντομα στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι σεβασμός του κράτους δικαίου απαιτεί ελεγκτικά εργαλεία και ενδεχομένως κυρώσεις που θα βασίζονται σε αρχές όπως η ανεξαρτησία, η μη πρόθεση τιμωρησίας ε, και η ανεξαρτησία. Αμεροληψία πρέπει να υπάρχει και να μην δοθεί πολιτική απόχρωση στις προσεγγίσεις. Η πρόταση του κανονισμού κινδυνεύει να αντιπροσωπεύει ε, το αντίθετο. Και πλήρω ημερίζομαι τις επικρίσεις που απίθυνε πάνω σε αυτό το ΔΕΚ. Παραθέτω κάποιε επικρίσεις. Ε, απόλυτη ε, διακρίση που γίνεται για την αξιολόγηση των ελλείψεων που υπάρχουν και παραβιάσεων που είναι μόνο στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά όλη τη διαδικασία. Και είναι απλώς θεατής παθητικός στο Κοινοβούλιο στην όλη διαδικασία. Οι πηγές αναφοράς και τα κριτήρια είναι σαφή για την αξιολόγηση την ποιοτική και η ιονή πλήρης έλλειψη εργαλείων αξιολόγησης. Όσον αφορά τις συνέπειες των μέτρων που υθετούνται, όσον αφορά τους τελικούς αποδέκτε των πόρων, δηλαδή τους πολίτε και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό, λόγω ελλείψεως, όπως λέει το ελεκτικό συνέδριο, λείπει και αρχική αξιολόγηση αντιχτύπου των μέτρων και υπάρχει και έλλειψη διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους κύκλους. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό να εξεταστεί και να βρεθούν εναλλακτικέ ε, προσεγγίσεις. Υποστηρίζω λοιπόν την απόπειρα του συναδέλφου Τέρι Κάμπρα να μεταφερθεί η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ορίων ε, των προαναφερθέντων ε, προαναφερθισών αρχών αναλογικότητας και έλλειψης πολιτικής απόχρωσης των προσεγγίσεων. Στην πρώτη φάση των εργασιών θέλω να εκφράσω ε, μια κάποια απορία και σύγχυση επί της ουσίας κυρίως όσον αφορά το βασικό δυστυχώ σημείο της νομοδοτήσεω. Ο προβληματισμός αφορά την αντικατάσταση της έννοια του κράτους δικαίου με κάτι πιο αφηρημένο σαν κριτήριο, των αξιών τη ενώσεω, αν και αναφέρεται στις αρχές του άρθρου 2 των συνθήκων. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, έννοιε όπως κράτο δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα ε, έχουν περιεχόμενο σαφέστατο σαφώς καθορισμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Όπως το Rule of Law Checklist της Επιτροπής της Βενετίας. Οι αξίες ε, αόριστα με αναφέρονται δεν έχουν αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα. Και αυτός ο χαρακτήρας των όρων αυτών όπως κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα όσον αφορά τη δυνατότητα απόδοσης δικαιοσύνης όσον αφορά τον, την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. Και είναι αβέβαιο ότι η έννοια αξίες έχει τη δυνατότητα να μπορεί κανείς να τη στηρίξει νομικά. Ίσως να μην υπάρχει καν νομική βάση για να εθετηθούν νομοθετικού περιεχομένου διατάξεις σχετικά με αυτή την έννοια. Ε, θα το συζητήσουμε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Μπάρμπαρα. Αυτά λοιπόν. Ο Σόμφωτ Απουσιάζει το ΕΛΚ. Στο σύνολό του σήμερα. Ο κύριος Ράντεφ μου έδωσε μακροσκελέστατη ομιλία προς ανάγνωση. Δεν θα δημιουργήσω το προηγούμενο και να διαβάζω δηλώσεις των μελών ακόμα και αν απουσιάζουν διότι θα καταλήξω να πρέπει να το ξανακάνω. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τι θα κάνω λοιπόν. Να πω ότι ήταν κάπως αρνητικός όσον αφορά την γνωμοδότησή σας και έχει διανύμει σε εσά τον εισηγητή και στους σκιώδεις την άποψή του και θα στενοχωρηθείτε πολύ από αυτά που θα είχε να σας πει. Θα χρειαζόμουν 7 λεπτά να τα διαβάσω. Δεν θα τα διαβάσω. Θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Γι' αυτό δεν το κάνω. Διότι θα ξαναβρεθώ σε αυτή τη θέση. Άρα δεν θα το κάνω σήμερα. Θα διανύμω στους σκιώδεις το κείμενο. Και θα δουν ποια είναι η σοφή άποψη του ΕΛΚ επ' αυτού. Αυτά λοιπόν. Άλλωστε, επ' αυτού, να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να απαντήσω εν συντομία σε κάποιες από τις παρεμβάσει που ακούσαμε και καλώ ορίζω επίσης με την παράταση της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί γιατί ενδεχομένω ε, να μας επιτρέψει να εξηγήσουμε σε κάποια μέλη της Επιτροπής τις βασικές αρχές της πρότασής μας. Το θέμα δεν είναι βασικά επικεντρωνόμαστε στην προστασία του προεπλογισμού της Ένωσης και αυτό προβλέπει το άρθρο 322 της συνθήκης και αυτή είναι η βάση οποιοδήποτε οριζόντιας νομοθεσίας για την περιορισμό των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί να επικεντρωθώ λίγο στο παιδί εφαρμογή, γιατί ακούσαμε διάφορες απόψεις εδώ, αποκλίνουσα στην Επιτροπή. Επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση με το κρατός δικαίου, γιατί το κρατός δικαίου αποτελεί μια σαφή έννοια, ορίζεται στο άρθρο της πρότασής μας, περιλαμβάνει την αρχή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της νομιμότητας, της μη αυθαιρεσίας, της απα... σωστής προστασίας των αρχών. Είναι σαφές λοιπόν ε, ποιες είναι αυτές οι αρχές και θα πρέπει αυτό να γίνει ξεκάθαρο ότι από τη μία μιλάμε για πολλές περιπτώσεις, δεν μιλάμε για μία και μόνη περίπτωση, αλλά παράλληλα ότι αυτό επηρεάζει και τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και η αξίωση της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε μέτρο προτείνεται θα πρέπει να είναι αναλογικός προς τον αντίκτυπο που έχει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να πω λοιπόν ότι δεν πρόκειται για κύρωση, πρόκειται για προϋπόθεση. Προϋπόθεση για χρηστή οικονομική διαχείριση. Αν σε κάποιο κράτος μέλος υπάρχει συστηματικά, γενικά, Ελλείψεις, υπάρχουν ελλείψεις σε, ένα από τους τομείς που αναφέρεται στο άρθρο 3. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σωστή δικαστική προστασία, δεν υπάρχει υπάρχει συστηματική παραβίαση των κανόνων για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πολύ απλά δεν έχουμε στην περίπτωση αυτή την ασφάλεια, τη βεβαιότητα ότι θα δαπανηθούν σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτή είναι η βάση της πρότασής μας. Η ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει κάποια γενική ρεσιμότητα για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο, γίνεται αποδεκτή από το δικαστήριο και σημαίνει ότι είναι διαφορετικές οι διαδικασίες και διαφορετικοί οι στόχοι από το άρθρο 7 της διαδικασία για τη συνθήκη. Εδώ λοιπόν προβλέπεται μια διαφορετική διαδικασία με διαφορετικό σκοπό δεν θέλουμε να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου ουσιαστικά κάθε αυτό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν είναι κύρωση, επαναλαμβάνω. Είναι προϋπόθεση για την ε, δαπάνη των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη με το άρθρο 7, ότι επικεντρωνόμαστε πολύ καλύτερα στην πρότασή μας αυτή για την σωστή και χρηστή οικονομική διαχείριση. Προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων. Να χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία για την τεκμηρίωση των πορισμάτων μας ε, στη διαδικασία σε αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχουν ε, αρκετές πηγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Επιτροπή της Βενετίας, εν μια σειρά εμπειρογνωμόνων και μπορούμε λοιπόν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουμε να μας διαφωτίσουν αν υπάρχει δυσκολία στην όλη διαδικασία. Τονίστηκε η ανάγκη να υπάρχει αμερομιληψία, να μην υπάρχει πολιτικοποίηση στη συζήτηση αυτή. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά και τα κράτη-μέλη επιτρέπει αυτή την αμερόληπτη διαμόρφωση, γιατί θα έχουμε την ε, ευκαιρία να κοιτάξουμε τα επιχειρήματα των κρατών μελών. Πάντα πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι τεκμηρωμένες. Αν καταλήξουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι διαφωνούμε με τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε και να τεκμηριώσουμε αυτή τη διαφωνία μας. Αυτή είναι η πρότασή μας λοιπόν προς το Συμβούλιο. Και φυσικά όλα αυτά υπόκεινται στην ε, στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είμαστε σε ένα ε, τέτοιο ένομο σύστημα και είμαστε υπόλογοι και στις αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τέλος, για την παρακολούθηση και στο δικαίωμα πρώτερης ε, διαβούλευσης. Αυτή η πρόταση δεν προέλθε από το πουθενά ήταν απόρρια τη συζήτηση για το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και είχαμε επίση και δύο αιτήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύο ξεκάθαρα ψηφίσματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ επίκαιρη και έγκαιρη και σωστή στη χρονική στιγμή αυτή η πρόταση για το επόμενο στη δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, και μα δείξατε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα προσέγεται για μια κλασική περίπτωση όπου ζητάμε συμβολή βάσει του άρθρου 54 σε κάτι τόσο θεμελιώδες για το πώς θα ακολουθήσουμε το θέμα του κράτους δικαίου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει λοιπόν ότι δεν πρόκειται για κύρωση, πρόκειται μάλλον για προϋπόθεση. Νομίζω ότι σε τελική ανάλυση με το αρθρό 54. Θέλουμε να δώσουμε και την ε, οπτική της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Αυτό και μόνο του θα έχει ένα πολιτικό βάρος. Θα μπορέσουν φυσικά και όλες και οι να διαβάσουν τα σχετικά σχόλια. Να μην υποτιμήσουμε όμως το γεγονός ότι θα υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και σε ό,τι αφορά το άρθρο 54 και από τον εισηγητή και από τους κοιόδες. Είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό. Όπως είπαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Συζητιέται εδώ και καιρό. Έχει ασφαλώς μεγάλο αντίκτυπο. Καλή τύχη σας εύχομαι. Τρέχει το θέμα αυτό. Σημαντική γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι που είσαστε λοιπόν εδώ και λυπάμαι που ήταν το τελευταίο θέμα αυτό θέμα μας αυτό πέμπτη μεσημέρι. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Τερικά Μπρας. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογίων είναι η 14η Νοεμβρίου. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ ποιητική συζήτηση. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επόμενη ποιοτικη συζητηση ευχαριστουμε την ευρωπαικη επιτροπη η επομενη συνεδρια θα λάβει χώρα στις 15 Νοεμβρίου 8.30 το πρωί στο Στρασβούργο. Και μετά 19 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.